Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Let us start our... Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση of each committee. της Επιτροπής Ήτρε. Σημείο υπαριθμών 7. Topic number 7. rules Κανόνες για χοντρική πώληση το, της ε, περιαγωγής. Η κυρία Κουπουλανάτρη είναι η συγγητρία. Η Ήτρε αντάλλαξε απόψεις για το θέμα αυτό στις 26 Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης που ετοίμασε η συνάδελφός μας. Σημαντικό θέμα, το γνωρίζουμε πολύ καλά, διότι θα καταργηθεί το τέλος περιαγωγής μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2017 στο βαθμό του δυνατού, κάτι που υποσχεθήκαμε στους πολίτες μας. Απ' την άλλη, επίσης, θα πρέπει να εξηγήσουμε και κάποια, να διαλύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις που υπάρχουν απροσδόκητες παρεξηγήσεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις συζητήσεις μας ακούγοντας την εισηγήτρια. Την κυρία Μιονπέτρα Κουμπουλανάτρη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μπορείτε να διαβάσετε την πρότασή μας. Ε, μερικά στοιχεία περιέχει. Πήρα κάποιες διαφάνειες για να δείτε εικονικά το στόχο της πρότασης. Βασίστηκα στο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρησιμοποίησε ε, συμβουλές συμβουλό, συμβούλων, έλαβε υπόψη τους στόχους μας και θα πρέπει να τροποποιηθεί η πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν επιτρέπει ανταγωνισμό στην αγορά λιανεμπορίου και χοντρικής περιαγωγής δεν επιτρέπει να πετύχουμε την κοινωνία του Gigabit, που είναι σημαντικότατο στόχο στην ψηφιακή στρατηγική και πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να στηρίξουμε τη χρήση δεδομένων. Και η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξασφαλίζει ότι οι καταναλωτέ θα μπορέσουν να έχουν ε, σχεδόν μηδενικά τέλη περιαγωγή και το ίδιο τέλο όπω στι χώρε του και ότι μέσω τη προτάσεω θέλουν να πετύχουμε τι καλύτερε τιμέ. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προωθεί αποδοτικέ επενδύσει ε, για μια ενιαία αγορά. για τη φωνητική τηλεφωνία πιστεύω εκεί ότι υπάρχει περιθώριο ανταγωνισμού και ανάκτησης του κόστους δεν αναφέρθηκα στο θέμα του SMS, είναι κληρονομιά αυτό. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω της χρήσης στοιχείων είναι πιο σημαντικά τα δεδομένα και από πολιτική σκοπιά και βλέποντας και τα ανώτατα όρια όσον αφορά την τιμολόγηση. Προτείνω να χρησιμοποιήσουμε πιο εύληπτα gigabit αντί megabit σαν μονάδα. Η πρόταση πρότεινε τη μέγιστη τιμή 8,5 ευρώ αναμονάδα για ένα γιγαμπίτ και θα κρατήσει αυτή τη τιμή μέχρι 6 χρόνια από τώρα. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο, η πρώτη εικόνα. Γιατί βάλαμε ανώτατα τα όρια. Διότι υπάρχει διαφορετική τιμολόγηση στα κράτη-μέλη. Και είδαμε ε, από τη συλλογή των στοιχείων ότι η τιμή επηρεάζει πολύ τη χρήση. Οι χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα αναμεγαμπίτ παρέχουν περισσότερη χρήση, μεγαλύτερη χρήση. Και οι χώρες με πιο υψηλό εισόδημα μεγαμπίτ καταλήγουν με τη μικρότερη χρήση. Η Φιλανδία έχει τη μεγαλύτερη χρήση, 5,5 γίγα το μήνα και η Ολλανδία 12 φορές λιγότερο και η τιμή στην Ολλανδία 15 φορές παραπάνω. Άρα θέλουν περισσότερη χρήση και χαμηλότερα εισοδήματα την εταιρεία ανά γίγαμπιτ. Όλες ε, οι εταιρείες είναι κερδοφόρες στη χώρα τους. Επόμενη εικόνα στην ίδια διαφάνεια επόμενο γράφημα. Βλέπουμε αύξηση πολύ μεγάλη παντού, πικίλη από 30 μέχρι 174% και η Λετωνία είναι η αλλαγή μεγαλύτερη. Αύξηση 174% στην ε, Λετωνία, διότι εκεί ε, θέσανε ότι δεν υπάρχει, αφαίρεσαν το όριο από τη χρήση ε, των δεδομένων. Το ίδιο στη Φιλανδία, στη Σουηδία προσφέρουν πακέτα με πολλά, με μεγάλο γκο ε, Στο Βέλγιο το όριο είναι 200 μέγα και όχι 5,5 γίγα. Βλέπετε μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών σε αυτή τη χρήση των δεδομένων. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανέλησαν τις διάφορες χώρες. Έγινε ανάλυση αναχώρα. Συνολικό κόστος για κάθε χώρα βλέπουμε. 8,5 βάλαμε εδώ. Δεν είναι καν στην κλίμακα είναι εκτός κλίμακας. Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι υπάρχει περιθώριο εμπορικών διαπραγματεύσεων. Δεν νομίζω ότι όλες οι εταιρείες αυτή την αγορά έχουν την ίδια ε, δυνατότητα διαπραγμάτευσης, την ίδια ισχύ και εξουσία και ξεκίνησα με πιο χαμηλό όριο, πολύ χαμηλότερο. Βλέπετε τι χρησιμοποίησε η Επιτροπή. Τέρα Consultants υπολόγισε το κόστος για την ε, χοντρική πώληση για την περιαγωγή και βλέπετε γιατί διάλεξα τα 5 ευρώ για να ξεκινήσω. Καλύπτει το κόστος χοντρικής περιαγωγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βλέπουμε την κατάσταση χώρες. Και μετά η νέα πρόταση για 4 ευρώ ε, καλύπτει όλα τα δεδομένα. Το ποσό δεν καθορίζει τα πάντα. Κοιτάξτε την άλλη άκρη του γραφήματος. πολλά κράτη-μέλη κατάφεραν με ένα ευρώ ή 1,5. Εστονία, Πολωνία, Ιρλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία. Ακόμα και η τιμή του ενός ευρώ μπορεί να καλύψει το κόστος της τιμής χονδρικής σε πολλές, πάρα πολλές χώρες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στα 8,5, στα 8,5. Πώς είχαμε τη διακύμαση του τιμών. Εγώ προτείνω σταδιακή μείωση. Δεν σταματάει η τεχνολογική εξέλιξη. Αυξάνεται η χρήση των δεδομένων. Χρειαζόμαστε νέα κλίμακα. Βλέπετε το γράφημα. Τι έχουμε ρυθμιζόμενες, ρυθμισμένες αγορές και ελεύθερες αγορές. Αν λέμε ότι μπορείς να... Αν θέλουμε να μην χρεώνεται ο πελάτης, θα πρέπει να το ρυθμίσουμε. Μια εταιρεία πληρώνει την άλλη εταιρεία. Πρέπει να ρυθμίσουμε ποιος πληρώνει ποιον και τι. Θα μειωθούν οι τιμές. Πόσο χρησιμοποιούμε τη λιανική τιμή. Η χοντρική τιμή αφορά εμπορικές συμφωνίες. Μπορεί να δει κανείς μετά όμως καλύτερα ποιες είναι οι τιμές λιανικής. Αν δούμε το Σεπτέμβριο, τιμές λιανικής, φέτος, πριν από κάποιους μήνες. Αυτά καλυφθήκαν με τις χαμηλότερε τιμές και η χονδρική είναι κανονικά ψηλότερη από τη λιανική. Άρα δεν είναι σωστή τιμολόγηση, βλέποντας την πραγματικότητα. Έχω αντίγραφο για σας. Δεν μπορώ εν συντομία να το παρουσιάσω. Είναι σημαντικό να το δείτε και να το διαβάσετε όμως αυτό αυτή Κάποιες εταιρείε πρέπει να πληρώσουν το μισό του το εισοδήματός τους σε άλλες εταιρείε. Και δεν είναι εύκολο αυτό. Πρόεδρε, κλείνοντας, το Συμβούλιο μπλοκάρει με αναστέλουσα ψηφία το όλο θέμα. Δεν είναι διαφορές μεταξύ κρατών μελών που μπορεί να δημιουργήσουν ανταγωνιστική αγορά. Και το θέμα είναι τι θα γίνει ε, μεταξύ των εταιριών και όχι μεταξύ κατώμελων. Σας, σας ευχαριστώ κύριος ε, Ρούμπικ από το ΕΛΚ. Να ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή. Νομίζω ότι ήταν ακριβέστατη η συγκήτρια σχετικά με τις χονδρικές όπως και τις λιανικές τιμολογήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να δράσουμε εάν είναι να έχουμε πρόοδο στο επίπεδο της ενιαίας αγοράς. Σε πολλά κράτη-μέλη ο ανταγωνισμός λειτουργεί πολύ καλά στο ιστορικό τους, αλλά έχουμε πολύ ακόμα δουλειά να κάνουμε στον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Και η τηλεφωνία δεν είναι το μόνο πεδίο στο οποίο έχουμε τέτοιου είδους ε, αποκλήσεις. Αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση ήταν ότι η αγορά τηλεπικοινωνιών στην ουσία γίνεται όλο και περισσότερο, όλο και ταχύτερα ψηφιακή ενιαία αγορά. Επομένω, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιών να υλοποιήσουν αυτό το άλμα προς την ψηφιακή τεχνολογία και να μπορούν να παρέχουν οικονομικές υπηρεσίες στους πελάτες τους και να πληρώνουν αξιοπρεπώς και τους εργαζόμενους τους. Νομίζω λοιπόν ότι η συνάδελφος ε, μας ε, παρουσίασε μια προσέγγιση ισορροπημένη και πλήρη. Τώρα, ο υπολογισμός σε gigabit ε, και όχι megabit ίσως για τους περισσότερους θα μπορούσε να είναι περίπλοκος Επομένως, ενδεχομένως η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν ίσως να μιλάμε για τα gigabyte σε ευρώ τελικά. Παρατήρησα πρόσφατα που ήμουν στην Ιαπωνία ότι ένα gigabyte, λέει ο μιλητής, μου στήχιζε 3 ευρώ στην πατρίδα ενώ στην Ιαπωνία 19.999 ευρώ ήθελαν να μου χρεώσουν, λέει ο μιλητής, δύο φορές το είπε, το νούμερο στην Ιαπωνία. 19.999. Άλλο ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι οι ε, virtual network operators γιατί ενδέχεται και με τα virtual network να έχουμε πρόβλημα. Κανονικά στο μέλλον αυτά θα πρέπει να έχουν μόνο εθνική τιμολόγηση. Γιατί οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τις καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Ο κύριος Τροσενόφσκι το PCR, παρακαλώ. Το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Κούμπουλα Νάτρη ε, για την παρουσίασή της και την πρότασή της και τον τρόπο τον οποίο κατάφερε να αναλύσει όλα αυτά τα δεδομένα κοιτώντας την παρουσίαση της διαφάνειας ε, κατανοεί κανείς αρκετά εύκολα ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, είτε μεταξύ βορρά-νότου, είτε μεταξύ και όμορων χωρών. Ε, το πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι ότι η πρόταση Μπέρεκ ε, θα ήταν αρκετά ακραία ενώ η πρόταση συγκήτριας είναι ακριβώς το άλλο άκρο. Ε, δυσκολεύομαι να φανταστώ πού θα ήταν ένα ενδιάμεσο, αν θέλετε, ισορροπημένο σημείο. Αν ήμασταν πιο φιλόδοξοι, δεν θα έπρεπε τελικά να μετακυλήσουμε ένα τμήμα του κόστους αυτό σε άλλες υπηρεσίες ή μήπως ε, θα απειλούσαμε και το σύνολο της αγοράς. Εγώ θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα αυτά που είχατε στην πρώτη τελευταία και την τελευταία διαφάνεια. Δηλαδή, πώς χρηματοδοτούν όλες αυτές τις υπηρεσίες οι φορείς, οι πάροχοι. Θα προτιμούσα εγώ να προχωρήσουμε επιφυλακτικά, με προσοχή, εν πάση περιπτώσει, ώστε να μην υπάρξουν αθέμητες συνέπειες, αθέμητος αντίκτυπος στην αγορά. Όμως, πραγματικά θεωρώ ότι η ανάλυση είναι πολύ καλή και μας προσφέρει ένα πλαίσιο για να μπορέσουμε να εξετάσουμε πώς θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Γιατί, επαναλαμβάνω, έχουμε δύο τελείως αντικρουόμενες ε, προτάσεις αυτή τη στιγμή και πρέπει να βρούμε μια ενδιάμεση θέση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Κούμπουλα Νάτρη. Είχαμε διάφορες επαφές και συναντήσεις και συζητήσεις για να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το όριο για τις ε, χονδρικές πωλήσει. Το σχέδιο είναι πολύ φιλόδοξο σχετικά με τα ανώτατα αυτά όρια. Επί της ουσίας πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τα όσα λέει η συγκήτρια Συνήθως βέβαια προτιμώ στους τριμερείς διαλόγους, στρατηγικά μιλώντας, να είμαι αρκετά επιθετικός. Αλλά έχουμε δύο μειοψήφια στο Κοινοβούλιο που επιθυμούν να μπλοκάρουν για διαφορετικούς λόγους. Δύο και όχι μία. Και δεν έχουμε χρόνο για τέτοια πράγματα. Διότι τα όρια αυτά είναι ουσιαστικότατα, απόλυτα αναγκαία για την τιμολόγηση του roaming, την πάυση του roaming από το 17. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα 8,5 και να φτάσουμε ταχύτατα στο επίπεδο που προτείνει η συγγετρία. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια συμφωνία. Χρειαζόμαστε τριμερή διάλογο. Δεν μπορούμε να μην έχουμε συμβαστική πρόταση, δεν γίνεται αυτό. Και το Άλντε προτείνει εμείς ως Κοινοβούλιο να ηγηθούμε προς την διερεύνηση αυτής της συμβαστικής πρότασης. Και προς αυτήν την κατεύθυνση θα κάνουμε και πρόταση τροπολογιών. Ευχαριστώ Ράιμοντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εμείς καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή έχει γίνει σωστή έρευνα, εξηγούνται τα πράγματα σωστά. Είναι σημαντική βάση για μια θέση του Κοινοβουλίου. Μπορούμε να συμφωνήσουμε βασικά με την έκθεση αυτή. Βασικό μας επιχείρημα είναι ότι θέλουμε να μειώσουμε το κόστος στο βαθμό του δυνατού για τον τελικό χρήστη. Αυτή πρέπει να είναι η θέση του Κοινοβουλίου, σκληρή θέση του Κοινοβουλίου. Δεν θα πρέπει να επιδιώξουμε εξ αρχής συμβιβαστικές λύσεις. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών σχημάτισε την εντύπωση ότι οι ομάδες ε, συμφωνούν και ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να μιλήσει σχεδόν με μία φωνή και αυτή είναι η προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε εν ώψη του τριμερούς διαλόγου για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό κόστος για το τελικό χρήστη. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μπορέλη, για το FTD. Συμφωνώ και εγώ όμως ευχαρίστησα τη συγγήτρια που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Πιστεύω ότι η ακολουθούμενη οδός είναι ορθή, προωθεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ όλων των επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων και πάνω απ' όλα καλύτερη υπηρεσία που παρέχεται στον πολίτη. Η πρώτης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την άποψή μου, δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. Εξετίμησα ιδιαίτερα την προσέγγιση τροπολογία 4 τη συντάκτρια που προβλέπει ετήσιε μειώσει για το μέγιστο τέλο τη περιεγωγή για τα δεδομένα. Θα ήταν εύκολο να φανταστεί ότι άμα το θέμα του roaming like at home θα αυξηθεί η κυκλοφορία, όγκος των ε, δεδομένο θα αυξηθεί. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα μέγιστο όριο αμετάβλητο για την επόμενη πενταετία. Υπάρχει περιθώριο και για μεγαλύτερε φιλοδοξίε και πιστεύω ότι σχετικά μπορώ να υποβάλω τροπολογίε που θα ακολουθήσω αυτή την κατεύθυνση. Και όσον αφορά την κυκλοφορία των δεδομένων και όσον αφορά και τι κλήσει. Πιστεύω, θεμελιώδε, ότι πρέπει να ενισχύσουμε και τη διαφάνεια πέρα από τον ανταγωνισμό προβλέποντας ε, και ε, κάποια μέτρα για τους εθνικούς φορείς. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε επί του λειτουργικού κόστους και θα πρέπει να... Ε, θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε καλύτερα το πάγιο κόστος, το overhead και το κόστος της ενεργοποίησης των υπηρεσιών roaming πρέπει να εξετάσουμε διότι χρησιμοποιείται αυτό σαν σκάνδαλο προβάσεις καταναλωτών το πάγιο στην Ιταλία μεγαλύτερες τηλεφωνικές εταιρείες σήμερα στο πρώτο λεπτό της κλήσης που γίνεται ή λαμβάνεται ή στο πρώτο SMS που αποστέλλεται ίσως ε, στο πρώτο megabyte που χρησιμοποιείται στο εξωτερικό ενεργοποιούν αυτομάτως για τους πελάτες χωρίς πρώτερη συνένεση ε, κατά αποκοπήν ποσά που δεν επιτρέπουν να πληρώνται σύμφωνα με την πραγματική καταναλωθή σε κυκλοφορία, αλλά ένα σταθερό κόστο που, που βγαίνει από 2 μέχρι 6 ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να ρυθμιστεί και να ελεγχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κιόρτσα έχει το λόγο. Για... Καλημέρα Πρόεδρε Τσόκα. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να χαιρετήσω την εισηγήτρια και όλους τους συναδέλφους και να πω σε όλους που χαίρομαι που μπορώ να συνεργαστώ μαζί στην Επιτροπή Ήτρε ως νεοαφιχθής δεχόμαστε θετικά τη βούληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επεξεργαστεί την πραγματική ανάγκη των πολιτών μας, των καταναλωτών μας και συμμεριζόμαστε το κριτήριο διασύνδεσης σταθερών συνδέσεων ε, μεταξύ το, της χώρας ε, και του, της εταιρεία από την οποία αγοράστηκε η ΣΥΜ. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα και θα προσπαθήσω να σας εκφράσω τον προβληματισμό μου. Πρώτα απ' όλα, είναι η πρώτη επίκριση του ΣΥΠΗΝ. Πρέπει να μπορούμε να αποφασίσουμε αν ένα χρήστης έχει δικαίωμα ή όχι να χρησιμοποιήσει το roaming like at home. Εκείνους τους εργαζόμενους που πηγαίνουν έρχονται σε άλλη χώρα καθημερινά. Άλλο πρόβλημα. Δεν είναι καθαρός ο μηχανισμός όσον αφορά τις ε, κυρώσεις για τους ε, χρήστες που δεν χρησιμοποιούν σωστά το roaming like at home μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα κίνδυνο. Να έχουμε υποκειμενική εφαρμογή της αρχής. Οπότε θα πρέπει και αυτό να ξεκαθαριστεί. Και όσον αφορά αυτά τα θέματα, επεξεργαζόμαστε σαν ομάδα τροπολογίες επικοδομητικού χαρακτήρα προς βελτίωση του κειμένου της Επιτροπής. Τελευταία σκέψη. Αυτά τα χρόνια είδαμε και άλλο στοιχείο, κάποιο πρόβλημα. Κάποιες εταιρείε μεταμόρφωσαν κάποιες ε, υπηρεσίες που παρήχαν από δωρεάν σε υπηρεσίες επιπληρωμή. Θα πρέπει να αποφύγουμε η προσπάθεια που καταβάλλεται για την περιαγωγή, το roaming like at home, να μην γίνει επιματέο όταν πετυχάνουμε αποτελέσματα θετικά για τον καταναλωτή, αλλά αυτό που γλιτώνει ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να καταβληθεί σαν συμπληρωματικό κόστο και να πληρώνουν από άλλη πλευρά το κόστος που γλιτώνουν οι καταναλωτέ μέσω άλλου κόστου που σχηματίζεται. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Άλλοι ομιλητέ. Δύο λεπτά μόνο, συνάδελφοι γιατί έχουμε πάνω από 10 ανθρώπους που στο κατάλογο. Η κυρία Δεκαστήγιο Βέρα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει κανείς καμιά αμφιβολία ότι για τη δέσμευση αυτού του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα και όλα στο, από τους βουλευτές αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ώστε <clears throat> να γίνει πραγματικότητα αυτή η κατάρρηση του roaming. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Οι προσπάθειες που έγιναν από πλευράς του Ευρωκοινοβουλίου για να πετύχουμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο πραγματικά ήταν εξαιρετικές προσπάθειες και ε, επετεύθη κάτι που απαιτούσε την ε, αναθεώρηση του πλαισίου όμως ε, που ήταν εύκολο να επιτευχθεί ουσιαστικά να αναζητηθεί δηλαδή μια οδός ενσωμάτωσης, ένταξης της πραγματικότητας των 28 εθνικών πραγματικότητων των αγορών που συναπατίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με τιμές, σε σχέση με συνήθειες καταναλωτικές, σε σχέση με τις ροές ε, από μία χώρα σε άλλη, αυτό δημιουργεί μία πραγματικότητα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου υπάρχει πολύ λίγος ο κοινός παρονομαστής, ο πανευρωπαϊκός. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτή την ε, ε, συνήθεια ή έδρασε μία, δύο, τρεις ή άλλες χώρες όμως ωστόσο είναι τόσο ευάλωτη αυτή η κατάσταση και υπάρχουν πάρα πολλές ε, τοπικές αγορές και όχι μια πανευρωπαϊκή αγορά. Αυτά όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εγώ ειλικρινά δεν γνωρίζω τα σχετικά με το, τις εκθέσεις. Γνωρίζω ότι έχει υποβάλει μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση ένα επιχείρημα μελέτης επιπτώσεων λέει. Αυτό είναι εκείνο το οποίο εγώ μπορώ σε αυτό να βασιστώ ειλικρινά. Πρέπει λοιπόν όμως να ληφθούν όλες αυτές οι πραγματικότητες υπόψη για να αναζητηθεί μια λύση. Γι' αυτό όπως ε, έγινε με τη ρήτρα της πιθανής κατάχρησης ή της ρήτρα για την αποφυγή, να αποφύγουμε απάτες, ε, ακριβώς ε, για αυτή την πραγματικότητα. Τώρα ήρθε η στιγμή να αναζητηθεί η λύση. Εγώ θα ήμουν υπέρμαχος περισσότερο του να ξεκινήσουμε με την πρόταση της Επιτροπής και να προσπαθήσουμε σε λογικές διορίες να επιτύχουμε μια αναθεώρηση των το, του κόστους προς τα κάτω σε σχέση με το 0,5 προς το 0,85 για παράδειγμα αναζήτηση μιας βιώσιμης λύσης που θα ξεκινά από την πρόταση της Επιτροπής αλλά και θα καταλήγει σε μια αναθεώρηση σε λογικές προθεσμίες των τιμών προς τα κάτω. Λόπες παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κανείς δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι είναι κατεπήγον να εγκριθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο για να μπορέσει να υλοποιήσει η Ευρώπη την υπόσχεση να καταργηθεί το roaming. Για να γίνει ανάμνηση του παρελθόντος το roaming δεν αξίζει να υιοθετηθεί οποιαδήποτε πρόταση. Πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις στα δίκτυα, να μην υπάρχει ε, οι, ε, χώρες που έχουν περισσότερο, περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές, να μην υποστούν ε, ε, ζημιές όσον αφορά το δίκτυό τους ή την ποιότητα των υπηρεσιών. Γι' αυτό αξιολογώ θετικά την πρόταση της Μία Πέτρα ως φιλόδοξη και με πρόθεση να επεξεργαστούμε την πρόταση της Επιτροπής για τις ανάγκες της αγοράς και την ανάγκη ενδεχόμενα να συνοδεύσουμε αυτές τις εκθέσεις με νομικές προτάσεις ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή ζημιογόνα επίπτωση. Ωστόσο, με ανησυχεί το ότι μεταξύ του προτύπου για το κόστος της Επιτροπής και των στοιχείων που αποκαλύφθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν από εθνικές ρυθμιστικές αρχές όπως της Ισπανίας, βρισκόμαστε σε υψηλότερα επίπεδα. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο που έχει μεγάλη εμβέλεια και τεράστια σπουδαιότητα σε ζώνες της ε, χώρας μου όπως για παράδειγμα η ε, χρονική στιγμή ε, που προξενεί πολλές φορές ε, και μια έκρηξη του κόστους και σε σχέση με το όσα έχουν συμπεριληφθεί στην αιτιολογική σκέψη 15 της πρότασης θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της αγοράς σίγουρα αλλά και οι επιστροφές των επενδύσεων στα δίκτυα για να διασφαλιστεί έγκαιρα η βελτίωσή τους. Ευχαριστώ. Μίστερ Μπόνι. Μπόνι παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Σκαμπουλανάτρη για την παρουσίασή της. Σε μια αναφορά για περαιτέρω συζητήσεις. Η έλλειψη ενωτά των ορίων για, για το χοντρεμπόδιο χοντρεμπόριο θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του κόστους για εταιρείε που θα είναι κάτι αρνητικό για τον εσωτερικό ανταγωνισμό και τις τιμές. Αυτό θα ισχύσει κυρίως για χώρες που στέλνουν κυκλοφορία περιαγωγής και για χώρες εκείνες για τις οποίες οι εγχώριες τιμές είναι χαμηλές και ωφελούνται ε, οι πελάτες από χαμηλές τιμές για όλες τις υπηρεσίες. Θα πρέπει τα όρια να καθοριστούν σε επίπεδο που επιτρέπει αποτελεσματική επίσκεψη των, ε, των δικτύων και ανάκτηση του κόστους. Έδειξε Μπέρεκ στη βαθμολόγηση που έκανα ότι η μέση τιμή σε ένα μεγαμπίτ, η τιμή αγοράς, εκεί συνεχώς μειώνεται. Ακόμα και όταν τα όρια χοντρικής παραμένουν αμετάβλητα. Είναι πολύ χαμηλότερα από τα ανώτατα όρια που θεσπίζονται, τρεις φορές χαμηλότερα. Η Ευρωπαϊκή της Επιτροπής δεν προβλέπει αναθεώρηση του επίπεδου των ορίων χοντρικής μέχρι 30 Ιουνίου του 2022. Ο καθορισμός των ορίων για την εξαετία αγνοεί τις τεράστιες μειώσεις τιμής μονάδας που αναμένονται τα επόμενα χρόνια σχετικά και με την εξέλιξη στην τεχνολογία πέμπτης γενιάς 5G. Θα πρέπει τα όρια να είναι πιο κοντά στις εκτιμήσεις του κόστου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πιο ισορροπημένη λύση και θα έτσι θα αποφεληθούμε από το roaming like home και δεν θα στρεβλώνεται ο εσωτερικός εγχώριος ανταγωνισμός. Θα επεξεργαστούμε δεόντως ε, τα διάφορα σημεία που ετέθησαν. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάλλας. Um, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω απολύτως με την ε, προσέγγιση της εισηγήτριας βήμα προς βήμα και να ξεκινήσουμε με τα πέντε έτη. Νομίζω ότι η, μεταρρύθμιση της αγοράς περιεγωγής ε, και στην χονδρική της ε, διάσταση είναι τμήμα της ίδιας δεσμίδας. Νομίζω ότι η Επιτροπή, μια και έχει υποβάλει την αρχική πρόταση, θα πρέπει να επανέλθει τώρα και στην ε, χονδρική αγορά. Αυτό δεν αφορά στη βιωσιμότητα των μοντέλων τιμολόγησης για τώρα ή για τρία ή για πέντε χρόνια, αλλά είναι η προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων στις ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα, περισσότερο όγκο δεδομένων κάθε μέρα. Και αυτό πρέπει να είναι απολύτως αντιληπτό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ με τις παρατηρήσεις ε, της συναδέλφου Μία Πέτρα και για όσους μιλούν για αύξηση από 1,5 στα 5 θα πω ότι το κόστος της χονδρικής είναι πολύ μικρότερο στα κρατημέλη αφενός, αφετέρου ίσως όλοι οι πάροχοι θα έπρεπε να δουν τα γραφήματα που παρουσίασε η συνάδελφος. Δεν θα έπρεπε να ε, αποσκοπούν στο μεγάλο κέρδος από λίγους πελάτες, αλλά στο μικρότερο σχετικά κέρδος από πολύ περισσότερους. δεν πρέπει να θεωρούμε τέτοιο είδους κατανάλωση ως είδος πολυτελείας σε καμία περίπτωση. Η εισηγήτρια δεν μας έδειξε στην, ε, στις διαφάνειες τι μπορούμε να αγοράσουμε με 30 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. Νομίζω ότι ε, στη Ρουμανία για ακριβώς την ίδια τιμή αγοράζει κανείς 6 GB ας πούμε όπως και στη Γερμανία. Ρουμανία και Γερμανία. Και έχουμε Deutsche Telekom και στη μία χώρα και στην άλλη από αυτές τις δύο. Και έχουμε και άλλους παραχούς στη Ρουμανία, την Orange και άλλους μικρότερους. Οπωσδήποτε όμως η, η καταναλωτική ισχύς είναι μικρότερη στη Ρουμανία από ό,τι στη Γερμανία, για να το θέσω έτσι με μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι η λογική, το ο λογικός μέσος όρος θα ήταν να πάμε στα 5 γιατί έτσι θα καλύπτονταν όλοι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντορίνιο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την εξαιρετική δουλειά που έκανε η συγγήτρια. Και επίσης να υπογραμμίσω κάτι, ότι έχουμε εδώ μια σταθερή βάση με βάση αυτή την έκθεση. Έχουμε δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος είναι να καταφέρουμε να καταργηθεί το roaming στην προβλεπόμενη ημερομηνία και το δεύτερο να μην υπάρξει επιζήμια επίπτωση στον ανταγωνισμό στην κοινή αγορά που είναι, θα είναι ψηφιακή η αγορά ενιαία για να μην υπάρξουν στρεβλώσεις στις περιφερειακές και ε, τοπικές αγορές. Και γι' αυτό αυτό που αναφέρεται στο σκεπτικό ενέα είναι πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να επιτρέπει στους όσους επιχειρούν να αντισταθμίζουν το κόστος ε, συμπεριλαμβάνοντας και τα κοινά κόστη με αυτό διασφαλίζεται διασφαλίζονται κίνητρα για τις επενδύσεις. Και αυτές οι επενδύσεις είναι το κλειδί για, σε αυτό το οποίο αναζητούμε. Δηλαδή, σε σχέση με ένα σωστό πλαίσιο για το πλαίσιο αυτό το οποίο θα επιτρέπει τις υπηρεσίες σε ε, θετικές τιμές γιατί είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται αυτό. Έτσι υπογραμμίζω την τροπολογία που υποβάλλει στο σκεπτικό ένα εισηγήτρια και προτείνει ότι σε σχέση με τους παρόχους θα πρέπει να αξιολογείται ετήσια και από την Επιτροπή αυτό. Πέρα από αυτά, αυτές οι εκθέσεις θα πρέπει να οδηγούν στο να αποφύγουμε στρεβλώσεις. Και αν υπάρξουν κάποιες στρεβλώσεις θα πρέπει να προτείνονται μέτρα επανόρθωσης. Θα καταθέσω μια τροπολογία σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Βιρκούνεν, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την παρουσίασή της, την κυρία Κομπουλανάτρη. Όταν ξεκίνησε η όλη προσπάθεια με την περιεγωγή, εδώ και πολλά χρόνια, ίσως να εστιαζόταν το Κοινοβούλιο στις τηλεφωνικές κλήσεις και στα σύντομα μηνύματα SMS. Όπως γνωρίζουμε όμως, συζήτηση για κινητή κυκλοφορία δεδομένων αυξάνεται τάχιστα. 60 με 100% κάθε χρόνο αυξάνεται η κυκλοφορία και θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη όταν προσπαθούμε να θεσπίσουμε και να ρυθμίσουμε την τιμή χονδρική. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε του καταναλωτέ σε όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιούν επίση και τα κινητά αυτά δεδομένα και αυτέ τι υπηρεσίε. Θέλουμε να έχουμε καλέ ψηφιακέ υπηρεσίε με κερδοφόρε τιμέ και αποτελεσματική αγορά σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας περισσότερο στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν πολλά δεδομένα. Το συζητήσαμε εκτενώς. Το θέμα του Roam Like at Home σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διάφορα κράτη-μέλη, διότι οι πελάτες χρησιμοποιούν κινητές υπηρεσίες ποικίλο τρόπο. Και όπως προανέφερα, είμαι Φιλανδή. Και οι Φιλανδοί πελάτες χρησιμοποιούν πάρα πολύ δεδομένα. Είναι οι πιο δραστήριοι χρήστες για δεδομένα σε όλο τον κόσμο. Στην κινητή τηλεφωνία Άρα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για, τους, ε, για τις εταιρείες μας, για τους παρόχους μας. Ε, θα πρέπει να μειωθεί, να το όριο για τη χοντρική. Αναφέρθηκε ότι το σχέδιο εκθέσεως Κομπουλανάτρη ήταν πολύ φιλόδοξο, αλλά αν δούμε τον όγκο των στοιχείων από πλευράς Φιλανδίας, τα όρια, τα ανώτατα χονδρική θα πρέπει να μειωθούν πολύ περισσότερο από αυτά που αναφέρονται στο σχέδιο εκθέσεως. Μπορούμε να βρούμε γι' αυτό λύση. Είναι σημαντικό όμως όλοι οι πελάτες και όλοι οι πελάτες στην Ευρώπη να ωφεληθούν από το πακέτο περιαγωγής και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και να τους ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούν και τα δεδομένα μέσω κινητής τηλεφωνίας γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε μια ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Κοχλίτσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο. Θα ήθελα να αναφέρω τον Μύροσλαφ Ράνστορφ, τον συνάδελφο που απεβίωσε πρόσφατα και που ανέφερε αυτό το θέμα για πρώτη φορά. Αυτή τη στιγμή κάνουμε λόγο για την κατάργηση του roaming. Θέλω λοιπόν να αποτίσω φόρο τιμή στον συνάδελφο με αυτόν τον τρόπο. Κάνουμε λόγο για σαφή θέματα και η έκθεση είναι σαφής. Ένα πράγμα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη, ότι το roaming είναι εκείνο το οποίο σε όλες τις μεθοριακές περιοχές δημιουργούσε άνισες συνθήκες σε σχέση για παράδειγμα αν κάποιος είχε ένα σήμα σε ένα αεροδρόμιο πότε ήταν ένα γερμανικό ε, μήνυμα πιο φτηνό το ίδιο σε σχέση με τα τσεχοαυστριακά σύνορα και στην Τουρκία σε σχέση με το, τα SMS ελεύθερα χρέωσης. Το είδαμε αυτό επειδή είχαν ένα είδους πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμοζόταν. Πολλοί παρέχουν τέτοια ε, στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο προσφοράς και μάλιστα ελκυστικά και χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση. Πρέπει αυτά να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με ιδιαίτερη επιτυχία αυτή την έκθεση και όλοι να, να θυμόμαστε το συνάδελφο που έδωσε το ενακτήριο λάκτισμα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Χέλμερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, λέει κύριος Χέλμερ. Δεν διατείνομαι ότι είμαι παίων για τα θέματα τηλεπικοινωνιών. Θα είναι όμως θέμα αγορών και οικονομικών και από αυτά γνωρίζω Είχαμε κάποιο συνάδελφο που παραπονέθηκε ότι νέα τέλη εισαγόντουσαν σε παλαιότερα ελεύθερες ε, υπηρεσίες παροχής καθώς προσπαθούν οι εταιρείε ε, να αντισταθμίσουν τα έξοδά τους. Είναι βασικό όμως αυτό ως αρχή. Όταν ε, δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε ένα οικονομικό πάροχο να, να μπορέσει να αντισταθμίσει, θα αναζητήσει αλλού την δυνατότητα αντιστάθμισης και πολλές φορές ε, θα είχαμε ταχύτερη αύξηση τελών ή ε, βραδύτερη μείωση τους ε, μια και γίνεται αυτή η προσπάθεια εξέβρεση στοιχείων από το roaming. Για παράδειγμα, κάποιοι οι οποίοι ανήκουν στο jet set θα μπορούν να εξοικονομούν κονδύλια, ενώ απλοί πολίτες που δεν πηγαίνουν και στο εξωτερικό ή και πάνε σπάνια στο εξωτερικό θα ανακαλύψουν ότι πληρώνουν περισσότερα αυτό είναι κάτι αρνητικό και οπισθοδρομικό. Δίνει, παίρνει χρήματα από τους πιο φτωχούς και τα δίνει στους πιο πλούσιους. Είναι ένα τέλειο παράδειγμα, Πρόεδρε, πώς σε σχέση με τις παρεμβάσεις στις τιμές αυτό το οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν ελεύθερη αγορά συνήθως δημιουργεί χωρίς εξαιρέσεις περισσότερες ζημιές από ό,τι όφελος. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Connect, τον κύριο Βίλεν, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη για τη συζήτηση και όλος ιδιαίτερα στην εισηγήτρια για την έκθεσή της. Εκτιμούμε διάφορα στοιχεία της έκθεσης. Ένα από αυτά είναι ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται το θέμα η Επιτροπή αυτή. Με ταχύτητα. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, είναι επίγον το ζήτημα. Εκτιμούμε το ότι η συγγήτρια λαμβάνει υπόψη τα δύο βασικά θέματα. Δηλαδή, από τη μία πλευρά θέλουμε βιωσιμότητα για τους παρόχους υπηρεσιών της Λιανικής και ανάκτηση του κόστους κάλυψη του κόστους από εταιρείε που παρέχουν χονδρική πώληση του, της περιαγωγής. Προσπαθώντας να τετραγωνίσουμε τον λόγο κύκλο, υπάρχει δυνατότητα παρέκκλησης από τον κανονισμό για λόγους βιωσιμότητας και όχι για ανάκτηση και κάλυψη του κόστους. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα τιθέμενα όρια επιτρέπουν κάλυψη του κόστους από πλευράς των εμπλεκομένων παρόχων. Τρίτον, εκτιμούμε τον τρόπο με τον οποίο η συγγήτρια παρουσίασε τα διάφορα ζητήματα βάσει στοιχείων. Μόνο έτσι μπορούμε να συζητήσουμε βάσει στοιχείων για να ξεπεράσουμε τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν. Επιτρέψτε μου να εκφράσω κάποιες επιφυλάξεις εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, αν εστιαστούμε επί των στοιχείων περί κόστους, θα πρέπει να είναι πλήρη τα στοιχεία από τη στιγμή που είναι στη διάθεσή μας. Όχι το κόστος δικτύου που παρουσιάζεται στην οθόνη και στο γράφημα, αλλά και το κόστος διέλευσης που προστίθεται. Γι' αυτό συμπεράναμε για τη Μάλτα ότι το κόστος είναι 0,67 και όχι 0,47 cents. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ σημαντικές. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά σύνεση όσον αφορά τη λειτουργία, την απόλυτη ισχύ κάθε μοντέλου. Στο βαθμό του δυνατού είναι τέλειο και βάσει των στοιχείων που υπάρχουν. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι τα, τα όρια είναι όρια διαφύλαξης. πρέπει να λάβουμε υπόψη και το περιθώριο σφαλμάτων λόγω της αβεβαιότητας του εγχειρήματο. Εξού και η πρότασή μας όσον αφορά τα δεδομένα του 0,85 cents ανά gigabyte που εξασφαλίζει και το περιθώριο λάθους αυτό το ποσό. Τρίτον, για την πορεία που ακολουθείτε, την πτωτική βασιστήκαμε σε στοιχεία του 2015 με προβολή προς το 2017 με όλους τους προαναφερθέντες όρους, προχωρώντας χρονικά στο μέλλον. Έχουμε με την πεποίθηση ότι η μεγαλύτερη χρήση και τεχνολογία που αλλάζει θα μειώσει τις τιμές μονάδας, όμως δεν είναι απόλυτη η προβλεψιμότητα. Είναι πολύ περιορισμένη. Γι' αυτό προτείνουμε έναν αριθμό και το επανεξετάζουμε το ζήτημα μέσω ρήτρα αναθεώρησης. Κατανοούμε ότι τα θέματα των μειώσεων αυτών των σταθερών συζητούνται και εδώ και στο Συμβούλιο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τις τοτικές αυτές τάσεις να τις εξετάζουμε με προσοχή βάση στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη και την αβεβαιότητα των στοιχείων. Τι ούτω τρόπος προσπαθούμε να συμβάλλουμε στις συζητήσεις που θα είναι δυσχερείς και περίπλοκες. Κατανοούμε ότι ακούστηκαν κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την τακτική τοποθέτησή σας. Δεν είναι δική μας θέση να σχολιάσουμε. Σημειώνουμε και αυτό το θέμα. Κλείνοντας, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, η συγγήτρια. Αν θέλετε να απαντήσετε στις παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, οι γραφικές απεικονίσεις θα είναι στο ίντερνετ στην σελίδα της Επιτροπής. Είναι από την Τέρα, είναι από την Κομισιόν. Κάποια έχουν δημοσιευθεί ήδη, κάποια άλλα όχι. Αλλά είναι αναλύσεις επί της ε, τιμής λιανικής. Αυτό που δεν απάντησε καθόλου η Κομισιόν είναι πώς είναι δυνατόν η τιμή χονδρικής να είναι πολύ υψηλότερη από την τιμή λιανικής. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν ήδη σήμερα να συμβαίνει αυτό. Και να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής που ομολόγησε ότι υπάρχει περιθώριο καθόδου με τις τιμές που είχε υποβάλει η Κομισιόν. Επίσης να πω ότι η ρήτρα βιωσιμότητας ε, σημαίνει ότι ένας πάροχος δεν μπορεί να παρέχει roaming όπως οι τιμολογήσεις οι εσωτερικές, οι εθνικές, οι εγχώριες. Δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να λέει ότι ορίστε καλύπτω τη ρήτρα βιωσιμότητας αλλά δεν παρέχω roaming. Δηλαδή πρέπει για όλες τις εθνικές αγορές να είναι δυνατόν αυτό. Με ρώτησε κάποιος πόσα δεδομένα μπορείς να αγοράσεις με 30 ευρώ. Αλλά αυτό δεν το έχω πρόχειρο, αλλά σε αυτά που θα δημοσιευθούν, που θα ανέβουν, θα υπάρχει και αυτό. Ξέρουμε ότι είμαστε 120 φορές πιο ακριβοί από άλλες χώρες και είμαστε όλοι ανταγωνιστικοί. Επίσης, οι πιο αποτελεσματικοί πάροχοι πρέπει να καλύψουν το κόστος. Και πρόεδρε, εγώ είμαι απόλυτα έτοιμη να προχωρήσουμε στους τριμερείς διαλόγους, αλλά για παράδειγμα η Πολωνία έχει που ήταν στην ε, μειοψηφία άρνηση κυρίας είχε μεγαλύτερη τιμή εισόδου από χώρε που δεν ήταν. Επομένως, σας παρακαλώ όλους, δείτε τα σχετικά μεγέθη. Η προθεσμία είναι ήδη αύριο. Αύριο. Εγώ είμαι έτοιμη να σας δώσω τα εδωμένα σε όποιον ενδιαφέρεται. Θα είμαστε όμως απολύτως έτοιμοι να ψηφίσουμε 29 Νοεμβρίου για να ξεκινήσουμε με τους τριμερείς διαλόγους. Υπάρχει χρόνος. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Προθεσμία λοιπόν για τις τροπολογίες είναι 13 Οκτωβρίου αύριο. Και η ψηφοφορία στην Ήτρε στις 29 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ όλους τους ε, ε, σκιώδεις, ε, ευχαριστώ τους προηγούμενους εισηγητές και τους συμμετέχοντες στη συζήτηση, την Κομισιόν. Πάμε τώρα στην πρωτοβολία Cloud. Παρακαλώ τον εισηγητή Σαπχάουζεν. Έχετε το λόγο. Νομίζω ότι έχω πέντε λεπτά, Πρόεδρε. Δεν είναι έτσι. Πρόεδρε, το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Αφορά στο, μέλος, στο μέλλον με συγχωρείτε, των επιχειρήσεών μας, της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής, στις ηλεκτρονικές τεχνολογίες, ε, χιλιάδες, εκατομμύρια ίσως θέσεις απασχόλησης και επίσης της ίδιας της επιστημονικής εξέλιξης διότι η πληροφορική επί του υπολογιστικού νέφους ή του cloud για να συνεννοούμεθα είναι η σόρευση της περισσότερης γνώσης σχετικά με τις σχετικές τεχνικές και τεχνολογίες. Επομένως, πώς μπορούμε να βασιστούμε στα πλεονεκτήματα, στα ισχυρά σημεία που έχουμε ήδη στην Ευρώπη. Γιατί δεν είναι ότι μας λείπουν οι επιχειρήσεις, Έχουμε μια πρώτη επιχείρηση, την OVH, στο cloud. Έχουμε επιχειρήσεις που ασχολούνται με μικροεπεξεργαστές, που δεν έχει η Κίνα, για να αναφέρω αυτό το παράδειγμα. Δεν παράγει μικροεπεξεργαστές η Κίνα. Και έχουμε και επιχειρήσεις λογισμικού. Είμαστε επίσης η Ήπειρος η οποία γέννησε το Linux μου φαίνεται λοιπόν πολύ σημαντικό ότι αν επιθυμούμε να οικοδομήσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία δεδομένων και γνώσης ηλεκτρονικής, πρέπει να βασιστούμε στα ισχυρά μας σημεία, στα πλεονεκτήματά μας και δηλαδή στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ήμουν εξεπλάγην, εξεπλάγην που η δουλειά αυτή που μου ανατέθηκε ακούγοντας τις επιχειρήσεις αυτές που είναι ηγέτες στο πεδίο τους. Τη δουλειά αυτή λοιπόν που έκανα εγώ δεν την έκανε η Επιτροπή. Και η έρευνα που έκανα με διαφόρους παρόχους ε, ανοιχτής επιστημονικής γνώσης, κάποιοι υπεύθυνοι του Ινστιτούτου Παστέρ, ο επιστημονικός διευθυντής της πρώτης αεροναυπηγικής επιχείρησης στην Ευρώπη, έχοντας τους ακούσει, δεν έχω καθόλου την ίδια ερμηνεία του Open Science με αυτή που θα μπορούσε να έχει η Κομισιόν. Ανησυχώ λοιπόν. Πώς είναι δυνατόν η Κομισιόν να μην έχει συνομιλήσει με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, πώς είναι δυνατόν η Κομισιόν να μην έχει ακριβή απεικόνηση, εικόνα του θέματος αυτού μέσω παρόχων επιχειρήσεων που είναι πολύ γνωστοί. Πέρα από το χάρισμα και την προσωπική ικανότητα που μπορούν να έχουν διάφοροι συνάδελφοι της Κομισιόν, πρέπει να ξεφύγουμε από την ε, ε, ευρωπαϊκή ενδοσκόπηση και να μην μας απασχολεί μόνο το στρατηγικό λόμπινγκ αλλά να μας ενδιαφέρει η μελλοντική μας ικανότητα να είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες με τον κλάδο, με τις επιχειρήσεις που έχουμε. Και η Κομισιόν υπό την έννοια αυτή έκανε τραγικό σφάλμα στην έκθεσή της. Η Open Science είναι ανοιχτή στην ακαδημαϊκή συνεργασία και έρευνα. Ήδη υφίσταται. Η διαλειτουργικότητα ναι, είναι κάτι που πρέπει να επιτύχουμε, αλλά έχοντας ακούσει τους υπευθύνου ασφαλείας λογισμικού στη Γερμανία και στη Γαλλία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η διαλειτουργικότητα αυτή εξαρτάται και από τα εθνικά συστήματα που έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα και από την εθνική αριστεία εμπειρογνωμοσύνη. Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των εθνικών αγορών και της ενιαίας αγοράς. Ο υπολογισμός ε, high performance, η EDS, η DASO που φτιάχνει υποβρύχια πυρηνικά μεταξύ άλλων, Έχουμε μία αγορά, ασχολούμαστε με περιθωριακές αγορές και δεν ασχολούμαστε πλέον με αγορά 300 δισεκατομμυρίων όπως είναι η των μικροεπεξεργαστών. Ασχολούμαστε δηλαδή με πράγματα λανθασμένης κλίμακας. Πιστεύω λοιπόν, Πρόεδρε, ότι χρειάζεται μια επανάσταση στα δεδομένα που ανήκουν σε αυτόν που τα παρέχει. Που πρέπει να καταφέρνει αυτός που παρέχει τα δεδομένα να αντλεί και ένα όφελος, ένα κέρδος οικονομικό από την παροχή αυτή. Η έκθεσή μου είναι εξαιρετικά επικριτική ως προς την τοποθέτηση της Κομισιόν Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη στα γαλλικά και μπορείτε να την έχετε και στα αγγλικά και είναι η... Ε, τα πορίσματα των ερευνών που διεξήγαμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος, εκ μέρους του ΕΛΚ. Mr. Chairman, <clears throat> dear colleagues. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι απογοητευμένος απόλυτα με την έκθεση που υποβάλλεται από τον Ζαν Λούκος Είναι εκτός ε, πλαισίου της ε, προτινόμενης ανακοίνωσης. Αυτή η ανακοίνωση δεν είναι για την βιομηχανία ή ε, <clears throat> των ημιαγωγών και σε σχέση με την ε, ε, ε, ανάδειξη του, του software του ήπιου λογισμικού ως του πιο ασφαλούς για την Ευρώπη. Δεν συμφωνώ με την σύσταση να απορριφθεί απόλυτα πλήρως η ανακοίνωση της Επιτροπής. Θα συζητήσουμε λοιπόν το περιεχόμενο της προτινόμενης ανακοίνωσης. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να θέσουμε στο τραπέζι κάποια θεμελιώδη προβλήματα γιατί είναι τόσο σημαντική η καινοτομία για την Ευρώπη. Επειδή είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν τα νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την Ευρώπη όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία. Να δημιουργηθεί το σκηνικό και το τοπίο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Ένα νέο σύστημα χρειαζόμαστε είναι καθήκον μας να προσθέσουμε στις ε, εθνικές προσπάθειες και τις ε, κοινέ ευρωπαϊκές προσπάθειες για να αλλάξει το πλαίσιο της ευρωπαϊκής καινοτομίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το νέφος, ε, το υπολογιστικό cloud, με τις υποδομές που θα μας δώσουν στο τέλος τους καρπούς από την ευρωπαϊκή ανοιχτή επιστημονική προσέγγιση του cloud. Τι χρειαζόμαστε εδώ ουσιαστικά. Πρώτον, να αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα της, ε, των εξελίξεων στα μεγαδεδομένα big data, να δούμε επίσης ε, την ε, χρηματοδότηση μέσω των δημοσίων κονδυλίων για την έρευνα υπό ασφαλείς όρους και προϋποθέσεις με σεβασμό για τα δικαιώματα, των, τα πνευματικά δικαιώματα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε θετικά Δεύτερον, να αντιληφθούμε ότι ο ανοιχτός χαρακτήρας είναι η πρόσθετη αξία και όχι η απειλή σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στα επιστημονικά επίπεδα. Γνώση συν γνώση μπορεί να δώσει την γνώση με πρόσθετη αξία που έχει σημασία και είναι κλειδί για την ανάπτυξη μιας καλύτερης αναβαθμισμένης ζωής για τους πολίτες. Τρίτον, να κατανοήσουμε ότι τα στοιχεία, τα μεγαδεδομένα open massa δεν κινητοποιούνται σε σχέση με κάποια συμφέροντα. Πρέπει να ανοίξουμε αυτά τα στοιχεία για μας ως πολίτες, ως χρήστες, ως καταναλωτές, ως επιστήμονες. Χρειαζόμαστε κανόνες και κανονισμούς. Πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε και να εργαστούμε για αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς. Δεν συμφωνώ με την πρόταση όμως ότι ο κατακαιρματισμός των data, των δεδομένων, μπορεί να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα. Τέταρτον, να κατανοήσουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τις ευρωπαϊκές ε, επιστημονικές εξελίξεις, εκμεταλλευόμενοι και τον ορίζοντα 2020 με ταχύς διαδικασίες, ε, ταχύ, διαδικασίες ε, ώστε να μπορέσει να υπάρξει υποστήριξη όσον αφορά τις ε, πηγές για χρηματοδότηση από την Ευρώπη που θα διασφαλιστούν. Είναι ο μόνος τρόπος ε, να αποφύγουμε να εκμεταλλευτούν κάποιοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την έρευνα, όπως τονίζεται στο σχέδιο έκθεσης. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση το να αποφύγουμε, του να αποφύγουμε τον κίνδυνο με αυτόν τον τρόπο και της ευρωπαϊκής προσπάθειας επιστημονικού ε, νέφους Πόσα σημεία έχετε ακόμα. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε με μια πρόταση. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Κατανοώ πρόεδρε, κατανοώ. Έχουμε και εμείς κανόνες και κανονισμούς. Λοιπόν, παρακαλώ να ολοκληρώσετε, να αναφέρετε ένα σημείο, ένα σημείο, το πέντε έστω και να ολοκληρώσετε. Ακόμα και κατ' το μεσαίωνα η, επιστημο, η επιστήμη δημιουργώντας μέσω των πανεπιστημίων αυτή την ε, πρόσθετη αξία όπως ε, προτείνεται. Ευχαριστώ λοιπόν εισηγητά. Είμαι έτοιμος με τις τροπολογίες μου να βελτιώσω. Ευχαριστώ. SND. Νίκα παρακαλώ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω το ότι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάγκη να υπάρξει μια απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε αναμφίσιμα να υποστηριχθεί αυτή η πρωτοβουλία του ε, υπολογιστικού νέφους και σε σχέση με την κατανόηση της προστασίας δεδομένων είναι καλύτερο να υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία στην Ευρώπη αντί να ε, μετατεθεί αλλού και μετά να ε, εμείς να μικτηρίζουμε για αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερο για μας στο τέλος τέλος να δημιουργήσουμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία για αυτό το νέφος. Χρειάζεται η τεχνολογία, χρειάζονται επενδύσεις σε ευρύτατη βάση. Από την άλλη πλευρά η ταχύτατη διαβίβαση δεδομένων που θα είναι πραγματικότητα και επιπλέον θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε λόγο για υπολογιστές, super computers, που και αυτό πρέπει να είναι μια προτεραιότητα. Αν δούμε πόσοι από αυτούς υπάρχουν σήμερα παγκόσμια και πόσοι από αυτούς βρίσκονται στην Ευρώπη, ε, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ή ε, να δούμε αυτάρεσκα. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι προφανές. Ε, είναι πρόδειλο ότι χρειάζεται αυτή η πρωτοβουλία και να την υποστηρίξουμε και να την βελτιώσουμε. Είναι ε, οπωσδήποτε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα που αποστέλλεται ισχυρό μήνυμα ώστε η ψηφιακή ε, βιομηχανία να δημιουργήσει πλατφόρμες για την ε, διοίκηση και είναι πολύ πιο αποτελεσματικό αυτό το σύστημα και για τη λογιστική και οποιαδήποτε συστήματα όσον αφορά την κεντρική ε, έδραση του ε, νέφους, του cloud και της τεχνολογίας του, αντί να διασπαθίζουμε κονδύλια για πράγματα τα οποία είναι περιτά. Και πρέπει αυτό στην ευρωπαϊκή επικράτεια να δημιουργηθεί και να βρίσκεται υπό την άμεση εποπτεία των ε, ευρωπαϊκών οργάνων χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα ε, safe harbor. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια πρωτοβουλία την οποία σίγουρα θα υποστηρίξουμε διότι είναι ένα πολύ σχηρό μήνυμα για την ε, ευρωπαϊκή ε, τεχνολογία και τις επιχειρήσεις ε, τεχνολογίας και πληροφορικής και επιπλέον θα πρέπει και η τεχνολογία να μπορέσει να προαχθεί. Να μην βρεθεί η Ευρώπη να χωλαίνει στον τομέα αυτών των τεχνολογιών, στον έφος. Εκ μέρους της Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. ECR, ο κύριο Φόξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπόνι και τον κύριο Νίκα για τις παρεμβάσεις τους. Προσβλέπω στη συνεργασία μας. Είναι καθήκον μας ως Ευρωβουλευτές να εξετάσουμε προτάσεις και να ελέγχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε και την ευθύνη να εξετάσουμε τον αντίκτυπο των προτάσεων όπως ή εμπροκειμένο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τον έφος και να αξιολογήσουμε την αξία που έχει για τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο. Απογοητεύομαι διότι το κείμενο που υπέβαλε η δεν μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο διότι το κείμενο δεν επικεντρώνεται επί της ουσίας της ανακοινώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν προσφέρει στην Επιτροπή την ενδεδειγμένη βάση ε, για να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι είναι σαν να συνετ τάχθη ε, σαν ανακοινωθέν ε, του Εθνικού Μετώπου για επικείμενες εκλογές. Αναφέρονται ξένες ε, ολιγαρχίες ψηφιακές, προστατευτικός είναι ο τόνος της εκθέσεως. Υπερβολικά χρησιμοποιείται. Οι σκιώδεις καλά θα κάνουν να υποβάλουν ε, τροπολογίες για να διαγραφεί η, η όλη έκθεση και να την συντάξουμε εμείς από την αρχή. Τα σχόλιά μου τα αφιερώνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευπρόσδεκτη πρόταση. Καλωσορίζω να δημιουργηθεί αυτό το ευρωπαϊκό νέφος για τις επιστήμες. Θα είναι ασφαλό ε, στο περιβάλλον για την ερευνητική κοινότητα και θα υπάρχει και ανταλλαγή των ε, δεδομένων βάσει πρωτοβουλίες ορίζων 2020. Ευπρόσδεκτο αυτό, αλλά πρέπει να προστατεύονται ε, τα δεδομένα και να υπάρχει και επιμερισμός αυτών. Να υπάρχει ανταλλαγή αυτών. Είναι χωρίς σύνορα ψηφιακός κόσμος. Όταν βλέπουμε το θέμα των προδιαγραφών θα πρέπει να συνεργαστούμε με εταίρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Τούτου λεχθέντο, δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το ρόλο να καθορίσει διεθνεί προδιαγραφέ και πρότυπα. Επίση, αμφισβητώ κατά πόσο το σχέδιο κειμένου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει τι ανάγκε τη βιομηχανία. Με, την... με το υπολογιστικό νέφο πρέπει να ενισχύσουμε του ε, καινοτόμου ε, φορεί και θα πρέπει να προωθεί το όλο θέμα και η βιομηχανία και η ζήτηση αγοράς. Δεν θα πρέπει να επιλέγει τους νικητές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό άλλωστε. Λοιπόν, αμφισβητώ κατά πόσο η δημιουργία ευρωπαϊκών υποδομών δεδομένων είναι κάτι που ζήτησε ο κλάδος και αν όχι κατά πόσο αποτελεί καλύτερη χρήση των χρημάτων του Ευρωπαίου Φορολογωμένου. Πρόεδρε, αναβοσβήνει το σηματάκι εδώ στο χρονόμετρό σας, θα σιωπήσω και προσβέψω συνεργασία ε, με τους συναδέλφους για τροποποίηση του σχεδίου εκθέσεως. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τρία λεπτά είχατε στη διάθεσή σας. Έκανα λαθάκι. Ζητώ συγγνώμη. Απόλυτα έγκαιρα μιλήσατε. Κυρία Βαν Νούεν, εκ μέρους της ε, Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ θετική, λέει η κυρία Νιούβενχάουσεν. Συνήθω τα βλέπω τα πράγματα θετικά. Σε αυτή την περίπτωση όμως δύσκολο αυτό. Το μόνο θετικό που μπορώ να πω είναι ότι ο συγητής είναι ενθουσιώδης για το θέμα. Αλλά εκεί θα σταματήσω. Σήμερα το πρωί όταν συζητήσαμε την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας Είπα ότι δεν ζούμε σε μια εποχή αλλαγών, αλλά ζούμε μια αλλαγή εποχών. Έχαμε και έχουμε τόσες νέες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα ταυτοχρόνως. Είτε είναι της διάστατη εκτύπωση, το διαδίκτυο των πραγμάτων, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά έρχονται μαζί ταυτόχρονα και όλα αυτά συνεπάγονται ανταλλαγή δεδομένων, μεγάλου όγκου δεδομένων. θέλουμε να δράξουμε τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες θα πρέπει να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα. Άρα πρέπει να έχουμε την κβαντική τεχνολογία. Εντάξει, η ιδέα είναι καλή να έχουμε προγράμματα για ε, το υπολογιστικό νέφος, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες ε, υποδομές για το νέφος. Το μόνο που θα ήθελα να κάνω θα ήταν να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για όλα αυτά. Όχι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίε εμπλέκονται κατά πολύ, αλλά και για πολλέ μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον έφο ποικιλοτρόπω. Μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων. Αφήνουμε ανεκμετάλλευτες πολλές ευκαιρίες, πιστεύω τώρα. Και θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν νέα τεχνολογία στον έφος και ε, σε ατομικό επίπεδο οι πολίτες. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αυτές τις δυνατότητες. Χρειαζόμαστε αυτές τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για οικονομική ανάπτυξη που επιθυμούμε διακαώς. Για να καταστεί εφικτό αυτό θα πρέπει ο δημόσιος τομέας να διευκολύνει τη δημιουργία των καταλλήλων συνθήκων. Πρέπει να τονώσουμε τη ζήτηση, να εστιαστούμε επί διασυνδεσιμότητας. Όλοι θέλουμε την κοινωνία του Gigabit και αν μιλάμε για Gigabit, με τα χαράς να ήμουν και εγώ φανατική οπαδός του Gigabit. Very Ευχαριστώ την κυρία Νέιβεν Χόιζεν. Η κυρία Ματίας ε, από την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι σε σχέση με αυτό το ζήτημα, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι υπάρχει ανάγκη σε σχέση με την επιστημονική κοινότητα και την κοινότητα γνώσης για αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπολογιστών νέφους. Πιστεύω ότι υφίσταται και έχει διεκδικηθεί από την επιστημονική κοινότητα και από τις επιχειρήσεις. Και είναι μια ανάγκη που αντιμετωπίζουμε και κάνουμε λόγο για μία από τις περιφέρειες του κόσμου όπου η ανάπτυξη και της ε, γνώσης ε, έχει ρόλο κεντρικό σε όλα αυτά. Και έχει λοιπόν ε, σε σχέση με την διεθνή παραγωγή πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Έτσι δεν έχει νόημα να μην έχουμε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία γιατί η ανυπαρξία αυτής της ε, ε, πραγματικότητας δημιουργεί αυτά τα προβλήματα και για τη βιομηχανία και που μετεγκαθίσταται σε άλλους τομείς, μια και στην Ευρώπη υπάρχει κενό και κινητοποιούνται αλλού και οι ερευνητές και αυτό οδηγεί στο να πρέπει να ε, τοποθετηθούν σε άλλες χώρες και τοποθετηθούν τοποθετήσεις με πιο άμεση και πιο ασφαλεία το εγκατάσταση για την απασχόλησή τους. Γι' αυτό λοιπόν η ύπαρξη υπολογιστών υψηλής τεχνολογίας υποχρεώνει να χρησιμοποιηθούν ε, υποδομές μη ευρωπαϊκές που η χρήση τους, η χρήση τους ε, πολλές φορές, τη χρήση τους την αγνοούμε. Και αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και δεν διασφαλιστεί ένα σύνολο όρων και προϋποθέσεων δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σχέση για παράδειγμα για τη συγχρηματοδότηση, την ε, ε, ρύθμιση και τα θέματα τα οποία θα πρέπει να ε, έχουν ξεχωριστό χαρακτήρα και ιδιαίτερα δεν θα δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθούν οι διαφορετικές υποεξέλιξη δραστηριότητες αν δεν έχουμε όλα αυτά Λοιπόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υπάρξει αυτή η ανοιχτή δυνατότητα. Είναι μια ανάγκη αυτό. Μια ανάγκη να υπάρξει και μια υποδομή για ευρωπαϊκά δεδομένα που θα χρησιμοποιείται από ευρωπαϊκά κονδύλια όπως τον ορίζοντα 2020 και που θα δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε με κάθε τρόπο τα ωφέλη της επιστήμης σε σχέση με αυτά τα δεδομένα. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε άλλη γραμμή κίνησης εμείς. Και αυτή είναι μια διάσταση θεμελιώδους σημασία και μια παρατήρηση εδώ που αφήνω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για όλα αυτά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση και η διαβίβαση δεδομένων θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες της επιστημονικής κοινότητας για την, ε, και για την εκπαίδευση και για να διατεθούν επίσης και κονδύλια για την ε, κατάρτιση και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων θα διασφαλίζεται πάντα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές και διατάξεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύονται οι επιχειρήσεις και το δημόσιο όσον αφορά την ασφάλεια. Μια και θα χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια, θα πρέπει επίσης ε, σε σχέση με ε, την διαφύλαξη αυτών των στοιχείων να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία για τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, έχω ακόμα στον κατάλογο πέντε ομιλητές, η κυρία Κάλλας. Πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με εκπλήσει η έκθεση αυτή διότι αντιφάσκει σε πολλά επίπεδα, απορρίπτει την πρώτη κομισιόν αφενός, αλλά ζητάει πολλές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αφετέρου, συνέργειες μεταξύ των παραγωγών λογισμικού και ηλεκτρονικών συσκευών, ε, και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες εμπορικές στην ηλεκτρονική τεχνολογία. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί δεν υποστηρίζει ο εισηγητή την πρόταση κομισιόν ή άλλη αντίφαση. Είναι η υποστήριξη που δίνει ο εισηγητή στο Linux, στο λογισμικό, στο λειτουργικό σύστημα δηλαδή. Η επιτυχία του Linux είναι ότι είναι ένα ανοιχτό σύστημα. Ανοιχτού κώδικα παντού στον κόσμο οι χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξή του. Και αυτό έρχεται σε απόλυτη αντίφαση με την υπόλοιπη κατεύθυνση της νομοδότησης. Για την πρωτοβουλία της Κομισιόν είναι σημαντικό να εστιαστούμε στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των όσων έχουμε. Αντί στην προσπάθεια δημιουργίας νέων πραγμάτων. Για τη διαλειτουργικότητα και τη διαχρηστικότητα χρειαζόμαστε digital identity, ηλεκτρονικές υπογραφές, καθότι τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή είναι στη φάση της υλοποίησης όλων αυτών. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γκροσέτ, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, Σημερίζομαι την έκπληξη των συναδέλφων στην ανάγνωση αυτής της έκθεσης. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει το ρόλο που της πρέπει στη διαχείριση των επιστημονικών δομένων. Ο υπόλοιπος κόσμος ε, προχωρεί γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Τώρα, ε, το άρθρο 1 βασίζεται σε κάποιες λανθασμένες αναλύσεις ε, και λανθασμένη ερμηνεία του HPC στα αγγλικά, του High Performance calculation και επίσης ε, στη δυναμική της ίδιας της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας του κλάδου. Τώρα δεν θα απαριθμίσω όλα τα σημεία που μου φαίνονται περίεργα, αλλά στο σημείο 11 φαίνεται να συστήνουμε την εγκατάλειψη του HPC από το οποίο εξαρτάται η πραγματική οικονομία και υπέρ κάποιων άλλων μοντέλων που δεν φαίνονται επαρκώς όρημα αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνονται έτοιμα να μας δώσουν ένα πραγματικό οικονομικό εμπορικό αντίκτυπο. Φαίνεται να βασιζόμαστε λοιπόν σε συστάσεις σε πραγμάτων που θέλουμε, επιθυμούμε να κάνουμε. Δεν πρέπει να αποφύγουμε να έχουμε στο πλωστάσιό μας, στη φαρέτρα μας, τα την αριστεία και την εμπειρογνωμοσύνη ε, διαφόρων στοιχείων ε, ηλεκτρονικής επιστήμης. Εν πάση περιπτώσει εκπλήσωμαι την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπικ έχει το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, διότι πολύ καλά τα τοποθέτησε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα τον πραγματικό κόσμο τον ε, βλέπουμε απέναντι στον εικονικό κόσμο. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτόν τον εικονικό κόσμο και οι αλγόριθμοι καθορίζουν αυτή τη στιγμή το τι θα γίνει και πώς πρέπει να πορευθούμε στο cloud, στο νέφος, στο υπολογιστικό. Και αν θέλουμε να κινηθούμε σε αυτό τον νέφος και να το κατανοήσουμε, τότε χρειαζόμαστε στον ορίζοντα 2020 μια νέα πλατφόρμα μια πλατφόρμα για τον έφος όπου θα αρχίσουν οι νέοι να εξοικειώνονται με αυτόν τον κόσμο εγώ είμαι αναλφάβητος, αγράμματος σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορώ ούτε να προγραμματίσω, ούτε να κωδικοποιήσω, δεν κατανοώ καν τη γλώσσα των υπολογιστών. Περί αυτού όμως πρόκειται. Η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να εξοικειώνεται με τις δεξιότητες και ικανότητες για τον κόσμο του νέφους, του υπολογιστικού νέφους. Και εδώ να μπορούν αυτά τα δεδομένα να αυτοπροσδιορίζονται από μας ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιος ε, λόγος ε, να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο διότι από τη μορφή αυτών των δεδομένων και τις δομές τους μπορούμε να συναγάγουμε νέα συμπεράσματα. Περί αυτού πρόκειται εδώ. Με το ευρωπαϊκό επιστημονικό cloud να δώσουμε ένα υπόδειγμα, να είμαστε πρωτοπόροι, να δείξουμε ότι εμείς ως Ευρώπη είμαστε σε θέση να αναλύουμε τα δεδομένα μας, να τα δομούμε και να συναγάγουμε τα συμπεράσματα. Δεν θα χρειαζόμαστε τον άλλο κόσμο, τις άλλες χώρες. Είναι δική μας ικανότητα και αρμοδιότητα και πρέπει να το αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί γι' αυτό. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής. Η κυρία, η κυρία σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, η έκθεση αυτή βασίζεται σε ένα πρώτο εκτιμώντας που λέει ότι οι στόχοι της Κομισιόν θα πρέπει να ε, συνδυαστούν με τους στόχους των υπηρεσιών πληροφοριών της ΗΠΑ για να υπερασπιστούν όλα τα, όλες τις ε, ηλεκτρονικές πληροφορίες που έχουν ήδη στη διάθεσή του για να διατηρήσουν την ηγεσία τους. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση. Ο Γκόραν Μάρβιν, ε, ο υφιστάμενος, ε, ο τρέχον πρόεδρος, ήταν ο πρώην πρόεδρος της Μπέρεκ. Τι να σας πω, εάν είχαμε προβλέψει αυτό το χαρακτήρα πολιτικού μανιφέστου της έκθεσης αυτής, ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε τοποθετηθεί διαφορετικά. Πρέπει κανείς ε, να μπορέσει να φιλτράρει όλα αυτά τα μηνύματα και σλόγγαν, προκειμένου να φτάσει σε κάποιες πτυχές της έκθεσης που είναι, ε, έχουν, είναι αξιόλογες, έχουν σημασία εν πάση περιπτώσει αυτό που τελικώς πρέπει να κάνουμε με την έκθεση αυτή για τα ανοιχτά δεδομένα, ε, για την επιστημονική έρευνα, για το cloud. Υπάρχει ένα θέμα υποδομών. Πρέπει να έχουμε την ε, κρίσιμη μάζα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα ε, εμπρός ως Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γίνεται με το high speed computing. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα διαλειτουργικότητας και υπάρχει ένα θέμα κατακαιρματισμού. Αυτές είναι θεματικές που εδώ αναφέρονται και οι οποίες είναι σημαντικές για να φτάσουμε σε μια υψηλότητα της ποιότητας διαχείριση δεδομένων που είναι στις δυνατότητες του ευρωπαϊκού κλάδου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, ευχαριστώ, συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο θέλει το λόγο, δεν βλέπω. Άρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους της ΓΔ Connect ο κύριος Σκόρδας, Γενικός Διευθυντής, παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το σχέδιο αυτό έκθεσης, για την πρωτοβουλία του cloud. Πολύ λυπούμεθα ότι ζητάτε την απόρριψή της, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε πολλά κοινά σημεία. Τα big data είναι η πρώτη ύλη της οικονομίας και έχουν μεγάλη προστατευμένη αξία πολλές επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές και φορείς μόνο τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν ποιο είναι το πραγματικό δεδομένο των big data. Συμμεριζόμαστε τις αρνητικές επιπτώσεις από το να μην είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες αυτές και την τεχνολογία αυτή. Τα δεδομένα που παράγονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή συχνά, που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, παράγονται συχνά αλλού και συχνά οι σχετιζόμενες επιχειρήσεις μετακινούνται στο εξωτερικό, όπου το η σχετική υποδομή είναι ήδη διαθέσιμη σε σύγκριση με το εσωτερικό του ερωικού εδάφους. Η πρωτοβουλία ακριβώς σε αυτά τα σημεία αφορά. Είναι σαφές ότι το άνοιγμα της πρόσβασης πρέπει να ενέχει, να καλύπτει μια σειρά προϋποθέσεις για την πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να είμαστε όσο ανοιχτοί γίνεται και όσο κλειστοί χρειάζεται. Σχετικά με το δυναμικό HPC χρειαζόμαστε υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα, χρειαζόμαστε υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όχι μόνο για την ακαδημία, για την επιστήμη, αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα και για τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό ακριβώς λέγει η ανακοίνωση. Το HPC μας επιτρέπει να ερευνούμε με ποιότητα και ακρίβεια τεράστιους όγκους δεδομένων. Και είναι ένας παράγοντας κλειδής ανατομίας και ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Επιτρέπει ε, σε, σε ολόκληρους κλάδους να μετακινηθούν προς ευφιέστερες παραγωγές, ευφιέστερα πρότυπα παραγωγής, νέες εφαρμογές, πιο καινοτόμε και για να δώσω ένα μικρό παράδειγμα, λόγω των ε, προβολών HPC η αυτοκινηστική βιομηχανία έχει μειώσει τον μήνα, τους μήνες που χρειάζονται για να προετοιμάσει την παραγωγή νέων μοντέλων ενώ πολύ γρήγορα επίσης μπορούμε να εντοπίσουμε ε, γενετικές εξελίξεις ε, στο γενετικό κώδικα που αφορούν την καταπολέμηση του, του καρκίνου. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να μειώσουμε τις πιθανότητες της εμφάνισης μιας νόσου στα μωρά σε δύο γενετικούς παράγοντες μέσω της σχετικής αυτής έρευνας. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο ανταγωνιστικά χρονικά πλαίσια σε σχέση με αυτά που κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα και η Ιαπωνία. Κυρίως οι Ηνωμένε και η Ιαπωνία που αναπτύσσουν τα δικά τους οικοσυστήματα HPC. Στην πρωτοβουλία λοιπόν του Ευρωπαϊκού Cloud η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος HPC και για την ανάπτυξη επίσης, την ευρυντική ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού επεξεργαστή. Και όπως πολύ σωστά υπογραμμίζει η έκθεση, πρέπει να ε, επιτύχουμε κάποιες συνέργειες, όχι μόνο για την ε, κατασκευή υπερυπολογιστών, αλλά για την καλύτερη διαχείριση των big data και του cloud computing. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα στην Ευρώπη που να συνδυάζει τα περιφερειακά, το λογισμικό, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες με τις διασυνδέσεις με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ των, ε, της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά και της ανταγωνιστικότητας που πρέπει να έχουμε. Πρόκειται για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος και ενδιαφέροντος που αυτή τη στιγμή ε, στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επίσης συμμεριζόμαστε τη θέση σας ε, για την ε, κβαντική υπολογιστική, των οποίων οι εφαρμογές θα είναι πολύ σημαντικές Ήδη είχαμε μια ανακοίνωση για την αγορά 2020 άνω του 1 δισεκατομμυρίου με πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ανά έτος. Είναι η φιλοδοξία της Κομισιόν να διαρευνήσουμε και την κβαντική τεχνολογία με μια πρωτοβουλία flagship ε, μεγάλης κλίμακας και εύρους ώστε να, να επιταχύνουμε την ανάπτυξή της και τη χρησιμοποίησή της ε, από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο φορέα Περιμένουμε ενδιαφέρον τις δικές τοποθετήσεις επ' αυτών για να βοηθήσουμε και εμείς ώστε να εξερευνήσουμε και να συγκλίνουμε προς μια θετική έκθεση. For Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια σας. Ήσασταν απόλυτα σωστός στην τήρηση του χρόνου που σας διατέθη. Κύριε Σιγητά, τα τελικά σας σχόλια. Πόσο χρόνο έχω, Πρόεδρε? How much time? Τρία λεπτά για να συνοψίσετε. Θα απαντήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς τον τελευταίο μιλητή. Καμιά φορά έχω την εντύπωση, οι συνάδελφοί μου δεν διάβασαν την έκθεση και ότι η πραγματικότητα να βάλετε για αργότερα, διότι αυτή η έκθεση δεν είναι υποκειμενική, ούτε μεροληπτική, ούτε ιδεολογική, ούτε είναι Είναι καρπός ακροάσεων που διεξήχθησαν με παρουσία ειδικών στον τομέα και απλώς συμπεριλαμβάνει αυτό που μας είπαν οι απαΐοντες. Απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτιμώ να μιλήσω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά σε εκείνους που δεν εργάζονται και υποκρίνονται ότι μπορούν να δώσουν μαθήματα. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπογραμμίσω ότι το Big Data, τα μέγα δεδομένα, και επεξεργασία στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να λάβει χώρα πάνω μόνο αν ευρωπαϊκές εταιρείες θα ασχοληθούν με το θέμα και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς αύριο τα στοιχεία αυτά τα δεδομένα όπως είναι της Amazon ή οι αμερικανικές εταιρείες που συμμορφώνονται με το Patriot Act πώς θα εξασφαλίζονται θα ασφαλίζονται οι προσωπικές πληροφορίες και άλλες εάν δεν υπάρχει ευρωπαϊκό νέφος που από την αρχή θα ελέγχεται από ευρωπαϊκές εταιρείες. Είναι σημαντικοί και οι μικροεπεξεργαστές. Έχοντας ακούσει τους ανθρώπους ε, του STM και της ΑΒΑΗ ότι μπορεί να υπάρχει διαφυγή πληροφοριών μέσω μικροεπεξεργαστών, αυτών που έχουμε τώρα. Μπορεί να είναι μικροεπεξεργαστής κατασκευής διαφορετικής, μπορούμε να έχουμε θύρες που ανοίγουν και διαφυγή δεδομένων. Πρέπει να απαντήσει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά την προστασία δεδομένων των πολιτών. Η έκθεση Μπόντεν, η οποία συνετάχθη εδώ και εισακούστηκαν και εμπειρογνώμονες που είχαν εργαστεί για την Google και τη Microsoft, στην ακρόαση υπογράμμισαν τη σημασία της προστασίας των δεδομένων που είναι ανέφικτη σήμερα στα πλαίσια των αμερικανικών εταιριών. Όσον αφορά τον τους υπολογιστές ε, υψηλών αποδόσεων και την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, προφανώς ε, συμφωνώ. Προσέξτε όμως, εκείνοι που ηγούνται στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο και των υπηρεσιών δεν χρησιμοποιούν, είναι γαλλική εταιρεία, δεν χρησιμοποιούν τους υπολογιστές υψηλών επιδόσεων, τα HPC. Ακούστε τους. Ακούστε την ADS, ε, τους επιστημονικούς αρμοδίους. Είναι, αυτές, είναι παιχνιδάκι το αυτό που λέτε υπολογιστές υψηλής απόδοσης όταν πρέπει ε, όσον αφορά τα μεγάλα δεδομένα, αλλά και το Ινστιτούτο Παστέρο ακόμα κάνει διαδοχική επεξεργασία ε, των δεδομένων μέσω σειράς ε, κανονικών υπολογιστών. Είναι η Pasteur, η ADS και άλλες εταιρείε το κάνουν αυτό. Πρέπει να είμαστε σοβαροί συνάδελφοι. Είναι αφόρητο να ακούω αυτά που άκουσα. Τώρα, ο Πρόεδρος, σας παρακαλώ, κοιτάξτε, δεν ισχυρισμοί, απαντώ στους δικούς σας ισχυρισμούς. Ή την πραγματικότητα να βάλετε για αργότερα, Πρόεδρος. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Η συζήτηση σε αυτή την Επιτροπή να παραμείνει εντός θέματος. Δεν θέλουμε προσωπικές συζητήσεις και αντεγκλήσεις μεταξύ μελών. Στις συζητήσεις δεν άκουσα κάποια, κάποιον ισχυρισμό ότι κάποιο απευθύνεται σε εσά προσωπικά. Αφορούσε η συζήτηση το περιεχόμενο της προτάσεως ή της προτάσεώς σας. Σας παρακαλώ λοιπόν. Κατήστε την ίδια, τον ίδιο τόνο στις συζητήσεις. Και έχετε 30 δευτερόλεπτα τώρα πια στη διάθεσή σας. Μάλιστα, Πρόεδρε να πω απλώς ότι η επίθεση παρόλα αυτά ήταν ιδεολογικής φύσεως. Και η σκληρή πραγματικότητα ε, πρέπει να μας καθοδηγεί. Ακούσαμε τις πραγματικές επιρρήσεις. Τώρα τους κβαντικούς υπολογιστές. Στέφω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζω, υποθέτω, ότι ήδη υπάρχει υπολογιστής κβαντικός στον Καναδά. Τον αγόρασε η Google, η NASA τον αγόρασε δεν είναι ενδεχόμενο πιθανότητα, είναι μια πραγματικότητα. Μετά, όσον αφορά το καπάστη δυνατότητα, διακόπτει ο Πρόεδρος, σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι. Το χρονοδιάγραμμα προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 20 Οκτωβρίου, 12 ώρα το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Ήτρε τον Ιανουάριο του 2017 και στην Ολομέλεια θα αποφασίσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Πάμε στο επόμενο σημείο. Το 9. Τροποποιητική απόφαση για την υιοθέτηση του ερευνητικού προγράμματος του ερευνητικού φορέα για άνθρακα και χάλιβα και πολιετής κατευθυντήριες γραμμές για τον λόγο πρόγραμμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Το ερευνητικό ίδρυμα για το Χάλιβα και Άνθρακα, το Ταμείο δημιουργήθηκε από πόλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα όταν εξέπνευσε η συνθήκη το έτος 2002. Άρα προ 10 τετραετίες το Ταμείο δίνει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ πάνω κάτω το χρόνο για έρευνα και καινοτομία στον τομέα του χάλιβα και του άνθρακα. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι τρία τέταρτα πηγαίνουν στο χάλιβα και ένα τέταρτο στον άνθρακα. Η αναλογία είναι αυτή. Πολύ περισσότερα χρήματα πηγαίνουν για αποθεματικά και για έρευνα στον τομέα του χάλιβα. Μαζί με πόρους από, το, από τον ορίζοντα 2020, η χρηματοδότηση είναι κρισίμου σημασίας για την προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια οικονομία που εκπέμπει λίγο άνθρακα, αυξάνοντα ταυτόχρονα τον ενεργειακό μα εφοδιασμό και κάνοντα τη βιομηχανία μα ανταγωνιστική. Η χαλιβουργία είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα της χαλιβουργίας που αντιμετωπίζει και προβλήματα. Και μάλιστα λόγω ε, των προβλημάτων του κλίματος. Το Ταμείο συναθρίζει βιομηχανικού εταίρου, μικρομεσαίε επιχειρήσει, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπό λοιπόν τη προτάσεω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι κατανοώ εγώ την πρόταση αυτή, είναι να τροποποιηθεί η νομική βάση μετά την περιοδική αξιολόγηση των κανόνων διαχειρίσεως του Ταμείου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δύο βασικούς ε, στόχους. Πρώτος στόχος βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω απλουστευμένων κανόνων, κάτι παρόμοιο με τον ορίζοντα 2020 και τις σχετικές προσπάθειες. Δεύτερον, εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφανώς, με τη δέουσα διαφάνεια και βέβαια με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια έκθεση εκ μέρους της Επιτροπής Ήτρε. Το προτείνω, δεν είναι υπό την προσωπική μου την ιδιότητα. Το συζητώ το θέμα σαν πρόεδρος της Ήτρε. Δεν ήθελα να προδικάσω τη θέση της Επιτροπής. Ανέφερα διάφορα στοιχεία, γεγονότα που θεωρώ ότι έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Τρία όλο ιδιαίτερος και θα ήθελα να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τρία σημεία. Δεν έχω πιστεί απόλυτα ότι η ευθυγράμμιση με τους κανόνες του ορίζοντα 2020 απαιτούν τροποποίηση της νομικής βάσεως. αλλαγή τη νομικής βάσεως. Δεν είμαι σίγουρος. Παρακαλώ, απαντήστε σε αυτό. Δεύτερον, η πρόταση δημοσίευθηκε αρκετές εβδομάδες πριν τους οριζόντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ομάδων εμπειρογνωμόνων πριν επικαιροποιηθούν αυτοί οι κανόνες. Και η επικαιροποίηση των κανόνων ίσως να έχουν σοβαρές συνέπειες για την πρόταση αυτή. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται ένα ψήφισμα για τον έλεγχο του μητρού που έχει τα ονόματα των μελών των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι πεπισμένος ότι η έκθεση για το ερευνητικό αυτό ίδρυμα, ε, το ταμείο θα πρέπει να μην ε, να συζητείται αλλά να μην προδικάσει τα αποτελέσματα των ε, εργασιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απαντήσει στις ανησυχίες που σας εξήγησα, διότι εν γέννη συμφωνώ με την πρόταση αλλά ίσως να υπάρχουν και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες προς διευκρίνηση. Σκιώδης εισηγητές εκ μέρους των φιλελευθέρων, ο κύριος Τελίτσκα, ο οποίος έχει και το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας στο θέμα. Εγώ βρίσκω ικανοποιητικό το σχέδιο σε κάποιες στοιχείες και λιγότερο ικανοποιητικό σε κάποιες άλλες. Η χρησιμοποίηση των ε, πόρων είναι σε κάποια κράτη-μέλη αρκετά περιορισμένη. Ε, θα μπορούσε να επιχειρήσει κανείς μία εξέταση του γιατί έχουν έτσι τα πράγματα και να φτάσουμε σε μια ικανοποιητικότερη χρησιμοποίηση. Και οι μεταφορές προς την, υπό την έννοια αυτή είναι καλοδεχούμενη παρατήρηση. Αλλά οι διαδικασίες υπό τις οποίες μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση και εδώ πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δεν μιλούμε για χρησιμοποίηση από πλευράς μεγάλης κλίμακας, μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, οι διαδικασίες υποβολής χρειάζονται απλούστευση. Μόνο και μόνο το γεγονό ότι είναι περίπλοκες ε, και αυστηρές οι προϋποθέσεις ε, και μόνο στα αγγλικά, είναι ένας περιοριστικός ε, παράγοντας. Από εκεί πέρα η ευθυγράμμιση με τους κανόνες ε, ορίζοντα 2020 δεν είμαι βέβαιος ότι είναι η σωστή κατεύθυνση, η σωστή λύση. Και εγώ θα ε, διερευνούσα περισσότερο ε, την όποια δυνατότητα απλούστευσης θα είχαμε, ώστε η διαδικασία να είναι πιο εύπεπτη για τους ενδιαφερομένους. Τώρα βέβαια πάντα προσπαθούμε να διερευνήσουμε την δυνατότητα δημιουργίας ε, ε, ούτως επίν κλάστερς μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων ε, και καλώς έχει αυτό. Αλλά ως προς το διασυνοριακό στοιχείο, αρχή προς την οποία, την οποία προσυπογράφω χωρίς καμία αμφιβολία, αναφερόμαστε σε δύο συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, τομείς που τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον άνθρακα είναι αρκετά περιορισμένη εστίαση στα κράτη-μέλη. Υπό την έννοια αυτή το, η διασυνοριακή πτυχή ε, θα ήταν όχι αναγκαστικά προβληματική, αλλά κάτι που θα έπρεπε ε, να δούμε κατά πόσο είναι πραγματική προϋπόθεση. Έρεση. Και για κάποιους τομείς οικονομίας αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό από ότι για άλλους. Ε, τώρα η ισόρευση της εμπειρογνωμοσύνης ε, στις ομάδες εργασίας ε, ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει τύχει καλύτερης προσοχής, αλλά αυτά είναι περιφερειακά και δευτερεύοντα θέματα επί των οποίων δεν θα επέκλειε και να υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Όμως αυτά είναι κάποια αρχικά σχόλια, κάποιες αρχικές παρατηρήσεις που θα είχα. αλλά βλέπω ένα έλλειμμα στο να είναι περισσότερο φιλική προς το χρήστη αυτή η έκθεση και κυρίως εκεί εστιάζονται τους παρατηρήσεις μου. Μάλιστα ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων τώρα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι συνεργαστήκαμε σε σχέση με την επιστήμη και τις επιστημονικές έρευνες για το χάλιβα και τον άνθρακα. Ωστόσο, οι κανόνες και οι κανονισμοί είναι ανεδαφικοί πλέον και πρέπει να επικαιροποιηθούν. Εμείς οι πράσινοι επιθυμούμε περισσότερη διαφάνεια. Θέλουμε η ελεύθερη προσπελασιμότητα στα έγγραφα να διασφαλίζεται και σε σχέση και με τις συμβουλευτικές ομάδες σε σχέση με τις, ε, σε όσους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια μέσω συμβουλευτικών ομάδων. Από τη δημιουργία αυτού του ταμείου βελτιώθηκαν οι τεχνολογίες. Έχει πολυμορφοποιηθεί περισσότερο η ενέργεια και το οικονομικό τοπίο σε μεγάλο βαθμό μεταβλήθηκε. Οι βιομηχανίες χάλιβα και άνθρακα περνούν μια πολύ σε, μεγάλη σε βάθος ε, αναδόμηση εδώ μπορεί να παρέμβουμε, μπορούμε να παρέμβουμε ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις λόγω κλεισίματος ορυχείων και βιομηχανιών και χαλιβουργιών και θα πρέπει να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη πιο ασφαλών και καινοτόμων τεχνολογιών όσον αφορά αυτές τις βιομηχανίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από μικρό χρονικό διάστημα επετέχθη η Συμφωνία των Παρισίων και θα αρχίσει να ισχύει από τον επόμενο μήνα. Γι' αυτό η πολιτική μας και τα ερευνητικά ταμεία πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο τοπίο η προαγωγή του άνθρακα βρίσκεται σε καθαρή αντίφαση με αυτό το στόχο και θέλουμε να σταματήσει η εκμετάλλευση του άνθρακα. Αυτές είναι οι προτεραιότητες των Πρασίνων και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας. Επ' αυτού ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Εντάξει κύριε Σιλικιώτη έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρέπει να πω δυστυχώ η σκιώδη συγκίτρια τη ομάδα μα, η συνάδελφο Παλώμα Λόπε, ε, δεν μπορούσε να συμμετάσχει στη σημερινή συζήτηση. Βρίσκεται σε αποστολή του Κοινοβουλίου στην Κίνα. Γι' αυτό θα, θα ήθελα να εξηγήσω εκ μέρου τη την θέση τη ομάδα μα. Το Ταμείο Έρευνα Άστρα και Χάλιβα έχει αποδειχθεί ω ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον εξυγχρονισμό των δύο βιομηχανιών που αναφίβολα έχουν πληγεί από την φιλελευθερωποίηση του εμπορίου και την κατάργηση των κρατικών σχεδίων στήριξη. Ωστόσο, πρέπει να προσέξουμε καθώ το Ταμείο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση τη παραγωγικότητα των βιομηχανιών, αλλά μπορεί, αν χρησιμοποιηθεί με λαθασμένο τρόπο, να, να οδηγήσει μονάχα στη στήριξη του ιδιωτικού τομέα. Για εμά λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα βιώσιμα σχέδια στου τομεί του Άθρακα και του χάλιβα θα επιλέγονται με γνώμονα τα συμφέροντα και τι ανάγκε τη κοινωνία, σύμφωνα με τι πολιτικέ των κρατών μελών και δεν θα ενισχύουν τα ιδιωτικά συμφέροντα. Προ αυτήν την κατεύθυνση απαιτείται να αξιοποιήσουμε τα συνδικάτα και να διαβουλευόμαστε μαζί του κατά τη διαδικασία επιλογή των έργων. Επίση, πρέπει να εισαγάγουμε κριτήρια ώστε να διασφαλίσουμε πω τα κονδύλια που δίνονται θα στηρίζουν ιδιαίτερα τι περιοχέ που βρίσκονται σε διαδικασία αποβιομηχανοποίησης και ταλαρίζονται από ψηλά ποσοστά ενεργείας. Μόνο έτσι θα ενισχύσουμε την κινητήρια δύναμη της κοινωνικής ανάπτυξης. Ε, τέλος, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε πως τα έργα που λαμβάνουν δημόσια στήριξη και είναι βιώσιμα θα παραμείνουν ανοιχτά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε δραστηριότητες να επιδοτούνται κάποιες βιομηχανίες και μετά να κλείνουν, ιδιαίτερα όταν αυτές εξακολουθούν να, να είναι κερδοφόρες. Ε, το λέμε αυτό γιατί γνωρίζουμε, για παράδειγμα, όπως την περίπτωση της ΕΧΚΟΚΑ στην Ισπανία, η οποία έλαβε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από του ιδιοκτήτες της προς όφελος των ιδιωτικών ενεργειακών ολιγοπολίων. Αυτό αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα του τι πρέπει να αποφεύγεται στα μελλοντικά έργα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much, colleague. Any other request for the floor? Ευχαριστώ συνάδελφε. Ζητάει το λόγο, δεν βλέπω. Ρόμπερτ Μπουρμανί, επικεφαλής μονάδος, τμήματάρχης της Γενικής Διευθύνσεως για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ Πρόεδρε Μπούζεκ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας και ε, συνδέεται το όνομά σας με τη συμβουλή που δόθηκε στην όλη επιτροπή. Θα συνοψίσω τα όσα υπόθηκαν. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στη γραμματεία σας για το επεξηγηματικό υπόμνημα που ετοιμάστηκε, παρομοίως θα το είχαμε συντάξει και εμείς. Αυτό το υπόμνημα που ε, συνοδεύει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασικά, δεν αλλάζουμε το πεδίο εφαρμογής ή τους στόχους ε, του Ερευνητικού Ταμείου για τον Άνθρακα και το Χάλιβα, απλώς ε, έχουμε σχηματίσει κατευθυντήρες γραμμές προς την επίτευξη τριών στόχων βασικά. Αποδοτικότητα, διαφάνεια και συνέργεια είναι οι τρεις στόχοι. Να εξηγήσω για την αποδοτικότητα. Κοίταξε, από όταν είναι ξεχωριστό ανεξάρτητο πρόγραμμα Ακόμα ε, ε, συνάπτουμε τις δικές μας συμβάσεις για την έρευνα λόγω της νομικής αυτονομίας του Ταμείου. Δεν υπήρξε συνεργασία και χρήση των εργαλείων του ορίζοντα, του Horizon. Θέλαμε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα του Horizon 2020 κυρίως όσον αφορά τα συστήματα ε, ε, πληροφορικής υποστήριξης, ε, τις συμβάσεις και να διευκολύνουμε τη χρήση γνωστών κοινοτικών εργαλείων. Και Κάποιοι που συμμετέχουν στο Ταμείο μας συμμετέχουν και στα ερευνητικά προγράμματα για την ενέργεια, για τη βιομηχανία κλπ. Αυτό το θέμα της απόδοσης, αποδοτικότητας μετά τη διαφάνεια. Μας χρειάζεται αυτό παράλληλα με τη σύνταξη των νέων κατευθυντηρίων γραμμών περί ομάδων εμπειρογνωμόνων, διευκρινίζοντας περαιτέρω τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες κάποιων φορέων που έχουμε στο Ταμείο το Ερευνητικό και εξηγούνται άριστα αυτά στο επεξηγηματικό αυτό υπόμνημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε τι βουλευτικέ ομάδε από τη μία και από την άλλη πολλέ τεχνικέ ομάδε που λειτουργούν στον τομέα του άνθρακα και του χάλιβα. Το κάναμε αυτό στην τροπολογία της, στην αλλαγή της νομικής βάσης παράλληλα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Ένα πιο συγκεκριμένο σχόλιο, όπως είπε και ο κύριος Μπούζεκ, παρατήρησα ότι υπάρχουν δισταγμοί όσον αφορά την υλοποίηση από αυτή την πλευρά. Θα κωδικοποιηθούν όλα αυτά στους νέο, στο νέο εσωτερικό κανονισμό και για τις συμβουλευτικές ομάδες και για τις πολλές τεχνικές ομάδες. Αυτό θα είναι στη δεύτερη φάση, μετά την αλλαγή της νομικής βάσεως. Τέλος, Λίγα λόγια για τις συνέργειες. Πολύ συχνά μας τίθεται το ερώτημα πλευράς συναδέλφων αρμοδίων, κυρίως από τους βιομηχανικούς κύκλους, πώς μπορούν να συνεργαστούν ε, με άλλα προγράμματα σε μια, με έναν τρόπο φιλικό προς το χρήστη. Βασική ε, πτυχή, αν χρησιμοποιεί κανείς τα ίδια εργαλεία, όπως συμβάσεις, ε, συμφωνίες για τα κονσόρτσια κλπ, είναι πολύ πιο εύκολο να τους δίδουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες. Το λέω αυτό στο εξή πλαίσιο. Το σχέδιο προτάσεως που υπευλήθη έχει συζητηθεί με τους βιομηχανικούς κύκλους και του άνθρακα και του χάλιβα. Στο τέλος λοιπόν πρέπει να πω ότι έχουν συμφωνήσει λίγο πολύ με αυτά που προτείναμε ως τελικό αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα. Αποδοτικότητα, βελτίωση αυτής, διαφάνεια, εγγυήσει για τη διαφάνεια και συνέργειες με άλλα προγράμματα που ενδιαφέρουν αυτούς τους κύκλους της βιομηχανίας. Αυτά και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά της. Επιτρέψτε μου λοιπόν να προβώ σε κάποια σχόλια. Τρία σημεία ε, έθιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα της διαφάνειας, το θέμα των νέων διαδικαστικών κανόνων που θα μπορούσε να αφορά στο σύνολο των τροποποιήσεων στους διαδικαστικούς δηλαδή κανόνες των ε, ομάδων εμπειρογνωμόνων. Οι συνέργειες είναι πολύ σημαντικό θέμα, αυτό συζητήθηκε με τον κλάδο. Δηλαδή είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και πολύ κοντά στο ενδιαφέρον των χρηστών αλλά και των καταναλωτών. Και ίσως το πιο σημαντικό από τα θέματα, η αποτελεσματικότητα και ε, θυμίζω ότι το πρόγραμμα είναι το ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου για τον Άνθρακα και τον Χάλιβα. Αλλά μεταξύ των δύο αυτών η κλίμακα είναι 3 προς 1 υπέρ του Χάλιβα. Και κανείς δεν έχει διαφωνία ότι πρέπει να προασπίσουμε Ο άνθρακα είναι πολύ μικρό μέρο του ταμείου. Αποτελεσματικότητα λέει η Κομισιόν. Φαντάζομαι ότι κατά του όρου του μηνύματο efficiency και οι πράσινοι δεν θα μπορούσαν να έχουν κάτι να επικρίνουν. Και στα ενεργειακά θέματα πάντα λέμε απόδοση πρώτα, αποτελεσματικότητα δηλαδή, και μετά από μακρά παύση Ανανεώσιμε πηγέ ή οτιδήποτε άλλο. Α τακτοποιήσουμε λοιπόν τις προτεραιότητές μας και ελπίζω ότι και η Κομισιόν θα προετοιμάσει την ανακοίνωση γιατί είναι μια αναγκαία υποστήριξη για την Επιτροπή μας. Το θέμα της αποτελεσματικότητας ή της απόδοσης ε, είναι πολύ σημαντικό και δεν το αρνούμε. Εμείς ακούμε τα μηνύματά σας και σας παρακολουθούμε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τις τροπολογίες που θα υποβάλλετε 25 Οκτωβρίου στην Ήτρε. Μετά έχουμε την συνεδρία των συντονιστών, αλλά ήθελα πριν από αυτό να πω ότι αύριο ξεκινάμε όχι 9 και 10, όχι 9 και 4, 9. Γιατί πρέπει να ψηφίσουμε. 9 η ώρα, ακριβώς. Με τις κάρτες σας έτοιμες για την ψηφοφορία την ηλεκτρονική. Σε άλλη αίθουσα, στην 4Q2. Μην κάνετε λάθος. 4Q2 αύριο Ευχαριστώ για την απογευματινή συζήτηση. Θα σας δω αύριο. <laughs>